Ε, ε. Good morning everyone. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίασή μας. Καλωσορίζω τον κύριο Γουαλτιέρη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και τα μέλη και τον δύο επιτροπών, μια και πρόκειται για κοινή συνεδρίαση. Και παρακολουθούμε από κοινό αυτό το θέμα, το λεγόμενο της φορονομίας ταξόνομη. Φαντάζομαι μπορούμε να εγκρίνουμε την σε διάταξη. Να σε ευχαριστήσω καταρχήν θερμά για την αγαστή συνεργασία που είχαμε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο συνεισηγητές, τον κύριο Eckhout και την κυρία Πιετικάινεν. Μία ώρα δυστυχώ έχουμε προβλέψει για την εξέταση του σχεδίου έκθεσης ε, των δύο συνεισηγητών. Ε, που έχει και 123 τροπολογίες. Χαίρομαι ιδιαίτερος που συσπηρωθήκαμε οι δύο επιτροπές για να προωθήσουμε αυτό το θέμα που είναι τμήμα του πακέτου βιώσιμης ενέργειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να έχουμε ε, αθεκτικά μονοπάτια για να κατα καταφέρουμε με βιώσιμες πηγές ενέργειας να υλοποιήσουμε τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό και θα πρέπει να συνεργαστούν οι δύο επιτροπές, ΕΚΟΝ και ΕΜΒΙ για το θέμα αυτό και ελπίζω ότι χάρη στη στενή συνεργασία μας θα στείλουμε και χειρό μήνυμα στο Συμβούλιο. Και γι' αυτό προσβλέπουμε στη σημερινή συζήτηση του σχέδιου έκθεση. Να δώσω και το λόγο στον κύριο Γουαλτιέρη που θα μας κάνει και αυτός κάποιο πια εισαγωγικά σχόλια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά συμμετέχουμε στα πλαίσια του άρθρου 50 σε αυτή την κοινή συνεδρία των δύο επιτροπών για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Και μια και ο χρόνος είναι μετρημένος και θα έχουμε και ψηφοφορίες αργότερα στην ΕΚΟΝ, ας στηρίσουμε πιστά το χρονοδιάγραμμα και γι' αυτό θα πω από την υποβολή σχολείων για να κερδίσουμε χρόνο χρόνο και να δώσω κατευθείαν το λόγο στους συνεισηγητές. Σύρπα, Μπάς, παραείστε ευγενικοί. Πρώτα η Σύρπα. Ευχαριστώ. Ως συνεισηγήτρια, εκ μέρους ε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, για αυτό το θέμα, θα μπορούσα να ξεκινήσω εγώ. Καταρχήν, τι κάνουμε οι δύο συνεισηγητές. Να ευχαριστήσω πρώτα τον Μπάσεκ Κότ για την ασθενή συνεργασία που είχαμε. Γιατί χάρη σε αυτή καταφέραμε να εξομαλύνουμε κάποιες διαφορές μας. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει τελείως διαφορετική προσέγγιση ε, στι βιώσιμες επενδύσεις ε, σε αυτή τη συσταλτική φορονομία και ε, κατευθυγράμμιση με τα, με, με τα κριτήρια σύγκρισης, τα κριτήρια αναφοράς μάλιστα. Και αυτό φαίνεται και στην άλλη έκθεση. Η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υποβάλει αναφορές μόνο για τα θέματα των κλιματικών επιλογών και να αφήσει στη φορονομία τα θέματα των ε, φιλικών προς το περιβάλλον φορέων και το θέμα των ε, ε, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου με βάση τη Συμφωνία των Παρισιών. Ενώ η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν διαφορετική Εμεί είπαμε ότι θα πρέπει να αρχίσουμε την υποβολή εκθέσεων για όλα, για όλους τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, κυβερνητικούς αντικτύπους και των επενδυστικών εταιριών, ώστε και οι επενδυτικές εταιρείες, επενδυτικές επιχειρήσεις να έχουν την πληροφορία και να υπο να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια στην υποβολή αναφορών για τις επενδυτικές τους πολιτικές. Και αυτό φαίνεται στην έκθεσή μας και στους δείκτες, αλλά και στις άλλες εκθέσεις περί δημοσιοποίησης. Η ιδέα είναι στην ε, ταξονομία και στην ε, δημοσιοποίηση, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος ε, να αντικατοπτρίζεται από τους δείκτες, κάτι που σε μεγάλο βαθμό το έχουμε αναπτύξει και με τον ειδικό τομέα. Έχουμε το παγκόσμιο benchmarking και επίσης έχουμε το γνώσα το, την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, του το ΙΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Eurostat επίσης κάνει τη δική της δουλειά και στην πλατφόρμα παρακολούθηση κυκλικής οικονομίας επίσης γίνεται αυτή η εργασία. Εμείς θέλουμε ε, να συμπεριλάβουμε και να τα ολοκληρώσουμε όλα αυτά έχοντας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση συνδυάζοντας τα σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων και τη φορονομία, το ταξόνομι σε αυτούς τους ε, βασικούς δείκτες. Να δούμε καταρχήν ποια είναι η κατανάλωση, σπόρους, ε, ενέργεια και το νερό και ποιος είναι ο αντίκτυπος στο οικοσύστημα των εκπομπών, ξεχωρίζοντας το διοξίδιο του άνθρακα, τη βιοποικιλότητα, καθώς και το κριτήριο της έμεσης χρήσης γης. Γιατί τώρα αυτή η υποβολή εκθέσεων είναι τόσο σημαντική. Αν έχουμε τις εταιρείες που παράγουν φιλοπεριβαλλοντικά, προϊόντα, πράσινα προϊόντα ε, και τις επιφορτήσουμε με διατυπώσεις ε, είναι αντιπαραγωγικό. Δεν θα έπρεπε να έχουμε τέτοια υπερβολική επιβάρηση. Γιατί αν κάποιος ε, θέλει να είναι ε, φιλικός προς το περιβάλλον θα πρέπει να έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί τον αντίκτυπο προς το περιβάλλον. Δεύτερο σημείο. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε εύκολα τι εστί μόνο πράσινος, green only. Γιατί όπως έχουμε πολλές αποχρώσεις του γκρι, έχουμε και πολλές αποχρώσεις του πράσινου. Αν για παράδειγμα πάρουμε τον οικοδομικό κλάδο, τον κατασκευαστικό, Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα είδος σκυροδέματος ε, ε, ανάλογα με το ποσοστό που έχει είναι πράσινο προϊόν γιατί εξαρτάται πόσο πως οι πόροι χρησιμοποιούνται και τι διοξίδιο του άνθρακα εκπέμπεται. και τι είδου ανακύκλωση χρησιμοποιούμε. Αυτό καθορίζει το πόσο το σκυρόδεμα είναι φιλοπεριβαλλοντικό ή όχι. Οπότε αφήνει, αφήνουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα στις αγορές να ορίσουν τα κριτήρια αναφοράς, τα benchmarks για το πώς ε, τι εστί φιλικός προς το περιβάλλον. Αλλά βέβαια εδώ καλύπτουμε όλους τους τομείς και προβλέπουμε τη δυνατότητα να μπορέσουν οι τομείς να προχωρήσουν, να βαθμιστούν και να κάνουν πιο φιλοπεριβαλλοντικές πράσινες, δηλαδή δραστηριότητες. Οπότε υιοθετούμε και την περιβαλλοντική διάσταση στην προσέγγιση μας. Μια και είμαστε και Επιτροπή Περιβάλλοντος σε τελική ανάλυση. Αυτό φαίνεται και στο πεδίο εφαρμογή. Τώρα καλύπτει όλα, όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά και όλα τα ταμεία και την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους παρόχους δανείων, είχαμε πει κάποιους περιβαλλοντικούς δείκτες, κοινωνικούς, κυβερνητικούς, ολοκληρώστε λέει ο Πρόεδρος. Ναι, καταλαβαίνω ότι αυτά είναι τα πρότυπα που θα πρέπει να αναπτύξουμε στη συνέχεια. Και τέλος, για τις λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση της φορονομίας, του ταξόνομη. Ε, είναι σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία της βιοπικιλότητας που είναι ενισχυμένη μένει σε σχέση με την αρχική πρόταση. Αυτό και είμαι στη διάθεσή για να απαντήσω σε απορίες. Περνάμε στον δεύτερο τώρα συνεισηγητή, τον Μπάσεκ Χόουτ, που για πέντε λεπτά το πολύ έχει χρόνο ομιλία. Ξέροντας τον εαυτό μου, θα χρησιμοποιήσω το μερτικό μου. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που μπορούμε μαζί με την ΕΜΒΗ και την ΕΚΟΝ συνεργαστούμε και εγώ συμμετέχω στις δύο επιτροπές και είναι πάντα ένας λογικός συνδυασμός η ΕΚΟΝ και τα περιβαλλοντικά θέματα να προχωρούν χέρι με χέρι αφού μιλάμε περί πράσινης οικονομίας. So in this setting we are και χαίρομαι που σε αυτό το σχήμα συζητάμε μαζί τι πολύ καλή εξέλιξη. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Να ευχαριστήσω τους συνεισηγητή της ΣΥΡΠΑ που κινείται στα πλαίσια της ΕΝΒΗ. Έχουμε διαφορετικές θέσεις και είμαστε από διαφορετικές πολιτικές ομάδες, άρα δεν συμφωνούμε στα πάντα. Είχαμε κάποιες σκληρές συζητήσεις, αλλά η κοινή μας αυτή έκθεση πιστεύω δίνει μια γενική επισκόπηση σχετικά με την κατάσταση του Κοινοβουλίου. Και βλέπω και στη σχετική πολιτική συζήτηση. Ένα-δύο στοιχεία να αναφέρω που ανέφερε και η ΣΥΡΠΑ. Πρώτα απ' όλα, πολύ συχνά επικρίνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι για αλλαγή τώρα θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδα άρχισε να ανησυχεί, αλλά την ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανα την πρόταση. Υπάρχουν πολλές νομικές προτάσεις για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, αλλά τώρα θέτουμε αυτό το θέμα της ιεράρχησης. Ε, αυτή η ιεράρχηση ε, θα χρησιμοποιηθεί και στα, σε μελλοντικέ εφαρμογές, όταν θα υποβάλουν πολιτικές πράσινης ε, οικονομίας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύστημα ταξινόμησης και αν κινηθούμε σωστά θα έχουμε παγκόσμια πρότυπα που θα θεσπίσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ακούμε αντιδράσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας παρακολουθούν. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε την πρόταση, που η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την πράσινη και τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Βλέποντας τις προτάσεις, βλέπουμε ότι σε κάνα δύο ζητήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως ήταν πολύ προσεκτική. Και εμείς βάζουμε τον πύχη λίγο ψηλότερα. Το σημαντικότερο είναι τι προσπαθούμε να κάνουμε την πρόταση. Να έχουμε μια ιεράρχηση που παίρνει χρήματα, χρηματοδότηση από κακές επενδύσεις προς πράσινες επενδύσεις. Θα πρέπει να γίνονται σωστά οι πράσινες επενδύσεις, οπότε οποιαδήποτε ετικετοθεσία πράσινη στο μέλλον θα αφαιρά πράσινη ε, ε, χρηματοδότηση πραγματικά. Και λέμε εμείς ότι η οικονομία οικονομικέ δραστηριότητε θα πρέπει να κρίνονται ε, όσον αφορά τις συνολικές τους περιβαλλοντικές επιδόσεις. Και σε κάποιο επίπεδο υπάρχει ε, μία μη βιώσιμη επίδοση. Είναι πολύ σημαντικό. Ταξινομία. Λοιπόν, θα, δεν πρέπει να ανησυχούμε να σπράσουν τη αυτή την ε, έκθεση. Αυτό που δεν λέμε ότι ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνουν χρήματα σε συγκεκριμένο τομέα αποκλειστικά. Τι καθορίζουμε. Τον αντίκτυπο που έχει η οικονομική δραστηριότητα και όπως το κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπου μια οικονομική δραστηριότητα έχει θετικό αντίκτυπο στην επίδοση συγκεκριμένου δίκτυ όπως εκπομπές άνθρακα. Can be και αν μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις και να μειωθούν οι εκπομπές, τότε είσαι στην πράσινη πλευρά. Αλλά η οικονομική δραστηριότητα που οδηγεί σε πολύ υψηλή αύξηση εκπομπών διεξουδίου του ανθρακός βεβαίως, τότε θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι αυτή η επίδοση είναι μη βιώσιμη. Πρέπει να καθορίσουμε τις οικονομικές δραστηριότητε. Δηλαδή, κάθε είδους εταιρεία βεβαία μέσω πράσινων χρηματοδοτήσεως θα βοηθηθεί στη μετάβαση που πρέπει να κάνει προς πράσινη οικονομία, όπω είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό ώψη του 2050, όπου θέλουμε να έχουμε μηδέν άνθρακα και μια οικονομία ουδέτερη όσον αφορά τον άνθρακα. Θα πρέπει να υπάρχει βοήθεια η χρηματοδότηση τομέων προς αυτή την κατεύθυνση. Και βάσει των επιδόσεων κινούμεθα. Αλλά προσθέτουμε ότι δεν είναι μόνο κάτι που αφορά θετική επίδοση, αλλά ελπίζουμε και πού βρίσκεται αρνητική επίδοση. Διότι αυτό θα δώσει τα αναγκαία κίνητρα για μετακίνηση οικονομικών ροών. Κάτι που θέλουμε. Και είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που η ΣΥΡΠΑ και εγώ προσθέτουμε στο πεδίο εφαρμογής της προτάσεως. Πέραν αυτού πιστεύουμε ότι πρέπει να διευρυνθεί το πλαίσιο της προτάσεως. Να καλύπτουμε και ποιος θα εφαρμόσει όμως, αυτή η ταξονομία, πρέπει να είναι ευρύτερη ε, βάση εντός του οικονομικού τομέα. Οπότε διευρύνουμε λοιπόν το πεδίο και διευρύνουμε και το πεδίο γύρω από την ε, αποκάλυψη και ανακοινοποίηση στοιχείων. Πρέπει να διευκρινίσουμε τη στιγμή που γίνονται κάποια πράγματα, πρέπει να αποκαλύπτονται, να παρουσιάζονται. Αυτό ήταν το πεντάλεπτό μου. Θα σταματήσω εκεί για το θέμα της επαλήθευσης μπορούν να πέσουν ρόλο οι διάφοροι φορείς, η ASA ε, και θέλουμε και στο μέλλον ε, να έχουμε τη σωστή, ε, τη σωστή προσέγγιση για την επιτεύξη των στόχων. Κινούμεθα βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσβλέπω στη συζήτηση. Και έτσι θα δούμε τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε μέσω των τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ορίστε. Πάμε στους κοιόδης εισηγητές. Για δύο λεπτά ο καθένα σας παρακαλώ. Η κυρία Μποναφέη, πρώτα απ' όλα. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ χαιρετίζω με ευχαρίστηση το ότι η πολιτική συζήτηση επί της εκθέσεως γίνεται στα πλαίσια της Επιτροπής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Οικονομικών. Λοιπόν, τα θέματα του περιβάλλοντος και τα οικονομικά θέματα δεν είναι σαν αντίφαση. Αυτό δείχνει. Να ευχαριστήσω τους συνδέφους Άοκεν και Πιτικάινεν για την πλήρη αυτή έκθεση που παρουσιάστηκε να κάνω ένα βήμα προς τα πίσω. Η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καθοριστεί ένα πλαίσιο που διευκολύνει τις επενδύσεις βιώσιμες αντιπροσωπεύει ένα θεμελιώδες βήμα για τη μετάβαση και αλλαγή του, οικονο... προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα του οικολογικού μοντέλου. Ε, Εμεί θέλαμε να περιγράψουμε κάποια σημαντικά ε, πλαίσια κανονιστικά που αφορούν τη βιωσιμότητα, όπως το θέμα της κυκλικής οικονομίας που θέλαμε να εξετάσουμε και τις ε, ενεργειακές πολιτικές. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να ειδωθούν όχι μόνο σαν πολιτικές ε, περιβαλλοντικές, αλλά σε μια βάση βιομηχανικής πολιτικής που είναι βιώσιμη. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι για να περάσουμε από τις ε, προδιαγραφές στην υλοποίηση αυτών, μέσω των πολιτικών χρειάζονται επενδύσεις και πρέπει να καταλάβουμε σαφώς ε, πότε πηγαίνουν οι επενδύσεις σωστή κατεύθυνση. Πότε η επένδυση είναι βιώσιμη και χρειάζονται πάρα πολλοί οικονομικοί πόροι. Λοιπόν, χρειαζόμαστε να συμφωνήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τι δραστηριότητε οικονομικέ που μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι βιώσιμε και βάσει ποιων δικτών ή ποιων παραμέτρων μπορούμε να αξιολογήσουμε με το επίπεδο βιωσιμότητά του. Και αυτό μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και αύξηση των επενδυτικών ροών προ τι δραστηριότητε που έχουμε μεγάλη ανάγκη. Μέσω σωστή αντιπροσώπευση των, ε, των διαφόρων θετικών αποτελεσμάτων αλλά και των κινδύνων που αντιμετωπίζει μία επένδυση, που θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για απάντηση τη σωστή επένδυση που γίνεται τεκμηριωμένη και εκείνοι που κινούνται στην οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να κινηθούν προς τη βιωσιμότητα. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε σαν ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών τροπολογίες που στρέφονται προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και κινούμεθα προς το φιλόδοξο στόχο του κανονισμού μέσω ε, των διαστάσεων των περιβαλλοντικών και της διακυβέρνησης και κοινωνικός άξονας ε, που ε, όλα αυτά διέπουν οδηγούν προς την ε, γενική βιωσιμότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζεντίλε έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώ από τις τελευταίες σκέψεις που εξέφρασε η συνάδελφος η κυρία Μποναφέη. Ε, αυτή η συζήτησή μας και το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών μου δεν μπορεί να μακρύνει από μια ανάγνωση που συμπεριλαμβάνει την κοινωνική πρόκληση σε αυτή τη μετάβαση, την πολύ περίπλοκη και δύσκολη. Τα οικονομικά, τα χρηματοπιστωτικά πρέπει να είναι ένα σημαντικό εργαλείο εργαλείο για να εντοπίσουμε πάνω απ' όλα τα εργαλεία και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να συνοδεύσουμε αυτή τη μετάβαση. Και να στείλουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς τους Ευρωπαίους άντρες και γυναίκες, στιγμές που περνάμε, που είναι δύσκολες και πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα μιας Ευρώπης που δίνει προσοχή στους πολίτες, άντρες και γυναίκες, μέσω πολιτικής περιβαλλοντικής που έκανε σημαντικά βήματα αυτά τα χρόνια και να αναφερόμαστε σε χρηματοδότηση που δεν έχει σαν απότερο σκοπό τον πλούτο για τον επενδυτή, αλλά και μία σημαντική μετάβαση προς ποιοτική ζωή και βελτίωση του περιβάλλοντος. Ποιοτική ζωή για τους ανθρώπους και βελτίωση του περιβάλλοντος. Πρέπει να συνεργαστούμε για να πετύχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα, να βρούμε ένα σημείο ισορροπίας. Ισορροπίας μεταξύ πολιτικής προσπάθειας να στείλουμε ένα σημαντικό μήνυμα σε αυτή την ευαίσθητη φάση της πολιτικής συζητήσεως έναντι των συμφερόντων των πολιτών και απ' την άλλη να διαφυλάξουμε το τμήμα των ε, επιχειρήσεων που θέλει να αποδεχτεί αυτή την πρόκληση. Πρέπει να ε, τελικά να έχουμε στη διάθεσή μας οικονομικά μέσα που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Λούκε. Good morning and uh, thanks to the colleagues for... Καλημέρα. Και ευχαριστώ για τα σχόλια μέχρι στιγμής. Ε, μιλάω εκ μέρους του ε, σκιωδού ε, ε, ε, του ECR ε, και η Swinburne υποστηρίζουμε το έργο το οποίο έχει γίνει ως τώρα από την Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις τρεις προτάσεις που ακολούθησαν που περιλαμβάνει και αυτό το νομοθέτημα για την ταξινομία. Θα θέλαμε να εφιστήσουμε προσοχή ε, στο έργο το οποίο έχει γίνει ως τώρα και ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, συμφωνία με το πακέτο βιώσιμης ανάπτυξης. Τώρα όσον αφορά τις απατήσεις ε, ε, ε, δημοσιοποίησης πληροφοριών θα θέλαμε να αποφύγουμε την αλληλεπικάλυψη και απαιτήσει οι οποίε θα απομακρυνθούν από την ποιότητα των δεδομένων που μπορούν να προσφερθούν από αυτό το νομοθέτημα. Επίση, θέλουμε επίσης να εξετάσουμε το πρόστιμα σχετικά με τις εκπομπές και να υπάρχει μια αντίστοιχη μετάβαση, όπως επίσης και οι δύο κατηγορίες. Το ECR θέλει να εκμεταλλευτεί τις ε, αλλαγές στην αγορά που βλέπουμε σε αυτό το τομέα ήδη και να προσαρμόσει έναν λόγο στην νομοθεσία. Έχουμε επίσης κάποια βασικά σχόλια αρχικά. Θα θέλαμε να χαιρετήσουμε την λήψη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων φαίνεται λογικό με βάση τον ρόλο που παίζουν ε, στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερο διευκρίνηση με βάση τα όσα συζητήθηκαν ε, και σχετικά με το αν αυτό ισχύει για όλες τις υπηρεσίες Επίση, ε, ε, για παράδειγμα. Επίσης, ε, σημειώνουμε την αλλαγή που βλέπουμε στις, στα προϊόντα τα οποία πλέον θεωρούνται βιώσιμα και αυτό έχει να κάνει και με, την, και με το label αρνητικού αντικτύπου. Και τέλος χαιρετίζουμε τη συμπερίληψη δικτών ε, και τα ε, κριτήρια ε, screening, τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά για να γνωρίσουμε το σημαντικό έργο το οποίο έχει γίνει διεθνώς σε αυτό το τομέα και τα άλλα εργαλεία είτε έχουν κάνει ταξινομία είτε όχι τα οποία είναι διαθέσιμα στους, χρωματο... Ε, στους επενδυτές. Ε, όταν εξετάζουμε τώρα τα ε, πρότυπα δεν νομίζουμε ότι θα πρέπει να απορρίψουμε τις υπάρχουσες πρακτικές στις αγορές. Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία όπως και διαφάνεια σε αυτό το πλαίσιο. Και χαιρόμαστε που βλέπουμε όμως το άρθρο 14 την επιβεβαίωσε της ε, ανάγκης ε, να συμπεριλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει θα εξετάσουμε στις τροπολογίες μας. Ε, θα χαρούμε για την περαιτέρω συνεργασία και συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από την Άλντι η κυρία Βίρινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί εισηγητές, σας ευχαριστούμε ε, για το σχέδιο έκθεσης. Ε, Έχουμε επεξεργαστεί εκ μέρου των φιλελευθέρων ε, τους τρεις φακέλους, έχουμε μια, έχουμε γενικότερη εικόνα και ένα όραμα σχετικά με το ρόλο τον οποίο θα παίξει η ταξινομία. Ο ρόλος αυτός ε, θα αποτελέσει μια κοινή γλώσσα, ένα γλωσσάρι σχετικά με το τι είναι βιώσιμο και με αυτό δεν εννοώ ότι θα πρέπει να είναι ένας κατάλογος άκαμπτος από ορισμούς, αλλά ένας κατάλογος ο οποίος θα ορίζει το πώς μια δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη. Για να έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο ανοιχτό προς τις ε, κοινοτομίες σε έναν τομέα ο οποίος εξελίσσεται, εξελίσσεται ραγδαίως. Ε, δεν είναι αναγκαίο και επιθυμητό να έχουμε άλλη μία πρόταση ε, η οποία θα αφορά την ε, δημοσίευση πληροφοριών. Κάτι τέτοιο δεν είναι χρήσιμο. Σύντομα θα θέσουμε τις βάσεις για ένα βιώσιμο πλαίσιο το οποίο θα παρέχει την ε, στέρεα βάση για τις δεκαετίες οι οποίες θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κυρμπάντη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρότασή τη και θα ήθελα να δώσω έμφαση στο πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο συγκεκριμένο τομέα οι βιώσιμε ε, επενδύσει και τα χρηματοπιστωτικά. Και πάλι είδαμε ότι ο κόσμο αυξάνει, αύξησε φέτο τι ε, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρωπου για ε, κατά 2% αλλά και το 17 εμφάνισε τελικά αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οπότε θα είναι σημαντικό να κατευθύνουμε τις επενδύσεις που αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο ε, προς μια βιώσιμη οικονομία. Να τις κατευθύνουμε λοιπόν ε, προς μια πιο πράσινη κατεύθυνση. Και ε, σε αυτό το θέμα είμαι πιο επικριτικός απέναντι στην Επιτροπή. Κατανοώ ότι είναι αναγκαία η ταξινομία, είναι μια νομοθεσία η οποία όμως θα μπορούσε να είχε γίνει πριν από 10 χρόνια. Το επόμενο βήμα θα είναι τώρα να μην ορίσουμε απλά το τι είναι οι πράσινες επενδύσεις. Είναι αναγκαίο να κατευθύνουμε όλες τις επενδύσεις προς μια βιώσιμη ε, κατεύθυνση και πιστεύω ότι η έκθεση του 2014 και ε, η δεύτερη που ακολούθησε φέτος ε, τον Αύγουστο της Παγκόσμιας Επιτροπής ε, για το κλίμα και την οικονομία δείχνει το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Επικεφαλής ε, της ομάδας αυτή είναι πρώην πρόεδρος του Μεσικού και δείχνει ότι τρισεκατομμύρια επενδύσεις που θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια, εάν γίνουν με βιώσιμο τρόπο, τα ωφέλη θα είναι πολύ μεγαλύτερα από το αν συνεχίσουμε όπως πράταμε ως τώρα. Για μένα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος δεν είναι να πρασινίσουμε το 5% των ε, επενδύσεων, διότι εν τέλει ο στόχος θα είναι να πρασινίσουμε το 100% των επενδύσεων και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε. Και ε, οι εκθέσεις που ανέφερα στην αρχή το δείχνουν αυτό και το πόσο αναγκαίο είναι δεν αφορά το να το ε, ε, προωθήσουμε, να το αποδείξουμε. Θα πρέπει να γίνει με ε, τις πολιτικές μας, με την σύνδεση των δημόσιων επενδύσεων προς αυτή την πράσινη κατηγορία. Θα πρέπει και κλείνοντας να μην έχουμε μονάχα ταξινομία για τις πράσινες κατηγορίες αλλά και για τις καφέ κατηγορίες και να αναπτύξουμε με πολιτικέ που να σχετίζονται με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Παπαδημούλη, έχει το λόγο τώρα. κύρια Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω του δύο συνεισηγητέ, τον κύριο Εκάουτ και την κυρία Πέτη Κάινεν, παρά το ότι είναι φανερό ότι υπάρχουν και σοβαρέ διαφορέ μεταξύ του, Αυτό που μας παρουσίασαν ως μεταξύ του συνδυασμό, ε, το θεωρώ μια ικανοποιητική αφετηρία για τη συζήτησή μας. Ε, ε σκοπεύω να εργαστώ λαμβάνοντάς το ως βάση και να καταθέσω πολλές τροπολογίες ε, επιδιώκοντας να πρασινίσει περισσότερο, κύριε Κάουτ. Δηλαδή, να ενισχύσουμε επενδύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας που να ε, είναι φιλικές προς στο περιβάλλον, φιλικές προστίσεις, τοπικές κοινωνίες, να υπηρετήσουμε τους στόχους που έχει θέσει και ο ΙΕ για αυτά τα θέματα. Και η Ευρώπη πρέπει όχι απλώς να ακολουθεί τους στόχους του ΙΕ, αλλά να πρωτοπορεί στην υλοποίηση αυτών των στόχων. Να ενισχύουμε την λογοδοσία και την δημοκρατική λήψη ε, των ε, αποφάσεων. Και ε, νομίζω ότι οφείλουμε σαν Ευρω... Ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη στιγμή που η Κομισιόν έχει παρουσιάσει ένα κείμενο κάπως καλύτερο από αυτά στα οποία μας έχει συνηθίσει, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε ακόμη καλύτερο. Που σημαίνει μακριά από την επιρροή των λόμπις που θεωρούν ότι η Κομισιόν έχει γίνει πολύ πράσινη αυτό είναι η ανάγκη να τρέξουμε γρηγορότερα για να υπερασπιστούμε το περιβάλλον που νομίζω ότι πιέζει την Κομισιόν και εμείς που λογοδοτούμε στους Ευρωπαίους πολίτες οφείλουμε να πιέζουμε ακόμη περισσότερο γιατί είναι θέμα προστασίας του περιβάλλοντας, βιωσιμότητας της οικονομίας, προσαρμογής της σε και υπεράσπισε τελική ανάλυση του δημοσίου συμφέροντος. Ευχαριστώ. Thank you um, Μάλιστα, τώρα από τα υπόλοιπα μέλη. Ποιο θέλει το λόγο, κύριε Γκροστέτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όντω, το σχέδιο δράση για τη χρηματοδότηση τη βιώσιμη ανάπτυξη που προτάθηκε το περασμένο Μάρτιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια πολύ αξιέπαινη και θετική προσπάθεια, πολύ ευπρόσδεκτη και ε, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο ότι χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο για να κρίνουμε αν μια οικονομική δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη ή όχι. Ε, ήδη ακούσαμε πολλά από τους προλαλήσαντες. Να σας υπενθυμίσω κάτι πολύ επίκαιρο. Στη Γαλλία στα τέλη Νοεμβρίου στο Παρίσι είχαμε τη μέρα για τη χρηματοδότηση του κλίματος. Μια διεθνή εκδήλωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την βιώσιμη χρηματοδότηση. Τότε μια μικρή κυβερνητική οργάνωση, η Oxfam, δημοσίευσε μια έκθεση που επιπλήττει τις έξι σημαντικότερες ε, γαλλικές τράπεζες για το γεγονός ότι δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει στην COP21 το 2015 στο Παρίσι. Με βάση αυτή την έκθεση της Oxfam στη Γαλλία, οι τράπεζες για την περίοδο 2000 2017 έδωσαν 43 δισεκατομμύρια για τα ορυκτά καύσιμα και μόνο 12 δισεκατομμύρια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν τηρούνται λοιπόν οι δεσμεύσει ε, της COP21. Θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να μας σημειώσουμε πρόοδο και πιο γρήγορα και για τα δημόσια δημόσιες επενδύσεις, κρατικές επενδύσεις και για τη ρύθμιση, το κανονιστικό πλαίσιο. Ήδη υπάρχουν κάποιες πρόπτικες ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, έχουμε τη φορολογία ε, και την υποχρέωση των θεσμικών επενδυτών να δημοσιεύουν στοιχεία για τα κριτήρια της επιλογής που έκαναν για τις τοποθετήσεις, τις επενδύσεις τους, αλλά η πρόοδος είναι αργή, γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, στις επενδύσεις μεταξύ του τομέα, του τομέα κτίριων ή των οχημάτων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα ή την ανάπτυξη των ε, δικτύων ε, θερμότητας. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί θα πρέπει τα κράτη να σταματούν να επενδύουν τόσο πολλά στα τα καύσιμα, αλλά να αντιστρέψουμε αυτή την τάση και να επενδύουμε περισσότερε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ευχαριστώ κυρία Γιατερμάκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρόταση, να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρότασή της και να τονίσω ότι εδώ και καιρό βλέπουμε ότι οι επενδύσεις απομακρύνονται από τα ορυκτά καύσιμα και επικεντρώνονται προς πιο φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις και πράσινα προϊόντα φιλοπεριβαλλοντικά. Βέβαια, θα πρέπει και οι χρηματοπιστικές υπηρεσίες να ταχθούν υπέρ μιας βιώσιμης χρηματοδότησης. Πάντως, οι αγαθές προθέσεις της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν αρνητικές παρενέργειες. Για παράδειγμα, το θέμα της ταξινομίας αναφέρθηκε εδώ. Και οι ορισμοί ε, θα πρέπει να εδράζονται σε ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία. Δεν μπορούν να υιοθετήσουν αόριστο τους ε, γενικούς ορισμούς. Σε ό,τι αφορά την ε, βιώσιμη διακυβέρνηση, ούτε και εκεί μπορούμε ουρανοκατέβατους ορισμούς να έχουμε και μάλιστα ε, ορισμούς που αν, αντιστρατεύονται οι φυστάμενες διατάξεις και ισχύουσα νομοθεσία. Θέλουμε ένα πλαίσιο βιώσιμη χρηματοδότησης που θα ρίνουμε όλους τους τομεί να είναι πιο στραμμένα προς το περιβάλλον οι επενδύσεις τους και επίσης και η στέγαση θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Ε, ε και κατοικίε γιατί είναι πολύ σημαντικό κλάδος. Ναι. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά, ο Πέτρο Σμιτ. Ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της ΟΚΕ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα μιλήσω γερμανικά, γιατί είναι πιο εύκολο να μιλήσω και να εκφραστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση. Είμαστε ε, από την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης ε, και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι η Επιτροπή ασχολείται με αυτό το θέμα. Όμως για εμάς δεν επαρκεί. Είναι πολύ λίγο. Έχουμε όλα τα στοιχεία, θα πρέπει να απομακρυνθούμε από μια οριζόντια οικονομία και να κατευθυνθούμε προς την ε, κυκλική. Χρειαζόμαστε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Οι αριθμοί της Επιτροπής το δείχνουν ξεκάθαρα. Χρειαζόμαστε επενδύσεις της τάξεως ε, του ενός δις ετησίως το λέει η Επιτροπή, το λέει η Ένωση Εργοδοτών της Γερμανίας ότι χρειαζόμαστε αυτές τις επενδύσεις και όταν βλέπουμε το προσχέδιο κάτι τέτοιο δεν επαρκεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν στο συνολικό πι δέλτα θα πει 40% συνολικά ποσό για να ε, το επιτέχουμε αυτό. Εδώ γίνεται μια συζήτηση όπου αναφερθήκαμε λιγάκι για αυτό σχετικά με την κοινωνική διάσταση. Δεν αφορά μονάχα την πράσινη διάσταση, αφορά και την κοινωνική διάσταση βλέπουμε στην Ευρώπη ότι στις εκλογές ε, οι ε, άνθρωποι, ε, οι πολίτες νιώθουν πιο αποκομμένοι, οπότε θα πρέπει και εδώ να υπάρξει βιώσιμη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση σχετικά με το ποια κατεύθυνση κατεύθυνση θα πάμε. Μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα η οποία αναφέρεται στον όγκο το πόσο παράγεται και όχι ε, η ποιότητα. Εάν λοιπόν αυτό το συμπεριλάβουμε και στην χρηματοδότηση θα βοηθηθεί και γι' αυτό το λόγο στο κείμενο το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή, αυτό δεν προχωρεί αρκετά. Επίσης, αρκετά από όσα υπόθηκαν ε, σήμερα είναι θέματα τα οποία υποστηρίζουμε και εμείς. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ο κ. Μπολτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η βιώσιμη οικονομία είναι βασική προτεραιότητα. Καλώς ορίζουμε τις προσπάθειες του Ευρωκοινοβουλίου να προχωρήσουμε γρήγορα στον τομέα, γιατί είναι σημαντικός. Η ταξινομία είναι ακρογωνίως λήθος του σχεδίου δράσεω για βιώσιμα οικονομικά. Με τα χαράς βλέπουμε ότι και οι δύο επιτροπές έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για τη μετώπιση του ζητήματος. Ε, τα βιώσιμα οικονομικά αφορούν να λαμβάνουμε πάντα υπόψη περιβαλλοντικούς στόχους στη λειτουργία του συστήματος και να προσαρμόζουμε δεόντως τις πολιτικές μας. Χρειάζεται να κινηθούμε γρήγορα. Είδαμε ανησυχητικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερε από ό,τι θεωρούσαμε. Οι συνομοθέτες ελπίζουν καταλήξουν συμφωνία επ' αυτού το ταχύτερο δυνατόν. Υπάρχει ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα, κυρίως για το κλίμα. Όπως ανέφερε ο συγκριτής Μπάς Εκχάουτ, έχει τη μεγάλη ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί στον τομέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προσπαθεί να πλησιάσει τους παγκόσμιους εταίρους μας και αυτούς που δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι, αλλά πρέπει να τους ταρακουνήσουμε όλους και να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Γι' αυτό η επίτευξη πολιτική συνένεση μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου και γρήγορα θα είναι κρίσιμη σημασία. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να ηγηθούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται μερόνυχτα ολόκληρα και σκληρά για τα βιώσιμα οικονομικά. Έχουμε δημιουργήσει ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων για το θέμα αυτό που μας βοηθά να αναπτύξουμε το σύστημα ταξινόμησης, προχωρούμε στην κλιματολογική ταξινόμηση και τα αποτελέσματα των εργασιών θα είναι έτοιμα του χρόνου. Οπότε ελπίζουμε ότι θα έχουμε το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο έτοιμο όταν χρειάζεται. Τελικά σημειώσαμε δεόντως τις διάφορες τροπολογίες του Ευρωκοινοβουλίου και προσβλέπουμε σε συνεργασία με όλους τους ευρωβουλευτές, ούτως ώστε, να καταλήξουμε σε μια κατάλληλη συμφωνία, καινοτόμα συμφωνία με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, Λίκος Γκουαλτιέρη. Έχουμε κι άλλο ένα που θέλουμε στα πιστού ΚΑΤΣΤΙΑΙ. Συγγνώμη, συγγνώμη που έχασα το ΚΑΤΣΤΙΑΙ. Λέει κύριε Περέζ, κοιτάξτε, θα ασχοληθούμε το θέμα της ταξινόμησης ανεξάρτητα με το θέμα της αποκάλυψη στοιχείων, δημοσιοποίηση στοιχείων και της βαθμολόγηση. Χρειάζεται συνεκτική προσέγγιση. Πρέπει να κινηθούν παράλληλα δύο επιτροπέ. Και η Οικονομική Νοσματική Επιτροπή να κινηθεί κατάλληλα. Ανησυχώ για τους δείκτε, για την προοπτική για τους δείκτε. Η προσέγγιση μα ε, ε, δεν ελάμβανε υπόψη ω πτυχές του πακέτου. Οι βασικοί φορεί. Ε, δεν είναι παρόντες στη σημερινή συζήτηση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια γέφυρα μετάβασης για τη σωστή ταξινόμηση. Να γίνει πλήρης ταξινόμηση, full-fledged ταξόνομη. Και θα πρέπει γρήγορα να βρεθεί μια τοποθέτηση για τους δείκτες. Διαφορετικά, η αξιοποιητική εστία του Ευρωκοινοβουλίου θα είναι άκρος εύθραυστη. Σας ευχαριστώ. Και να ξαναδώσω το λόγο στους δύο συνεισηγητές για τα τελικά σχόλια. Η συρπαπητικά είναι. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Όντω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε προηγούμενες εκθέσει. έχει υπογραμμίσει τη σημασία που έχει η συνάφεια, η συνοχή μεταξύ των τριών εκθέσεων. Το επισήμαν όλε οι πολιτικέ ομάδε. Θα ήταν τραγικό διαφορετικέ νομοθετικέ προτάσει να ακολουθούν διαφορετικέ κατευθύνσει και να α, αντιτάσσονται η μία στην άλλη. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη συνοχή, τη συνάφεια μεταξύ αυτών των τριών νομοθετικών προτάσεων. Δεύτερον, θέλουμε στην πρόταση να εναρμονίσουμε τις υπάρχουσες πληροφορίες. Όχι να αλλάξουμε την ε, υφιστάμενη νομοθεσία. Και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ε, ξε, όρους για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τους επενδυτές και με βάση την παρούσα νομοθεσία και τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες να έχουμε ε, μια πρόταση που θα έχει αντίκτυπο παγκοσμίω, γιατί η χρηματοδότηση των αγορών είναι, γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και θέλουμε παγκόσμια πρότυπα λογιστικά. Οπότε θα πρέπει προηγουμένως ε, να δούμε και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες και πώς θα υποβάλουμε τις εκθέσεις. Ε, αυτός είναι ο στόχος του πακέτου ε, της βιώσιμης ε, χρηματοδότησης και της ταξινόμης ταξινομίας. Ευχαριστώ, ο κύριος Εκχότ. Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Να ευχαριστήσω απλώς τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους και τα σχόλιά τους. Έχω την αίσθηση πάντως ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και ξέρουμε ποια άγουσα θέλουμε να ακολουθήσουμε Θέλουμε απλώς να καταλήξουμε σε κατάλληλες συμβαστικές ε, τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι υπάρχει υποστήριξη για την ε, κατεύθυνσή μας. Επίσης, να τονίσουμε τη συνάφεια και τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πακέτων, να μην υπάρχουν ασυναρτησίες και σωστά τα σχόλια για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Είναι σαφές ότι αυτό που κάνουμε εδώ στο δικό μας ε, θέμα, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αντιβαίνει τα όσα αναφέρονται στη δημοσιοποίηση. Γιατί ε, στη δημοσιοποίηση στοιχείων και ταξινομία πρέπει να περιλαμβάνουμε και περιβαλλοντικά στοιχεία. Για πότε που δεν είναι περιλαμβάνουμε τα κριτήρια περιβάλλοντος κοινωνίας και διακυβέρνησης. Και σίγουρα θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε αντίφαση μεταξύ των διαφόρων νομοθετικών προτάσεων. Ούτε έχουμε ώρα να κατέβα τις προτάσεις, δεν επινοούμε τίποτα καινούριο. Απλώς λέμε ποια είναι, ε, ποιοι είναι οι στόχοι, μετριασμός των κλιμάτων, των κλιματικών αλλαγών, ε, κυκλική οικονομία, βιοποικιλότητα. Με βάση αυτό, αυτό θα κρίνονται οι επιδόσεις. Με βάση αυτά τα στοιχεία. Δεν υπάρχει τίποτα στοιχεία. Τίποτα καινούριο ε, αλλά θα δούμε πώς θα, με τι δείκτες θα, θα ε, ε, λαμβάνεται υπόψη η επίδοση και θα βαθμολογείται η επίδοση. Και για όλα αυτά συνεχίζει τις προσπάθειες και η Ευρωπαϊκή και είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Ε, με προβλημάτισε κάπως η αργή πρόοδο στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να πιέσουμε και το Συμβούλιο για να επιταχύνει τις εργασίες, γιατί ξέρουμε ότι είναι αρκετά ε, βραδικίνητες ε, και επίπονες οι διαπραγματεύσεις, επειδή έχουμε πολλές κατεξοδότηση πράξεις και οι μεγαλύτερες χώρες δημιουργούν κάποια προβλήματα στο Συμβούλιο και χρονοτριβούν. Πάντως θα πρέπει να επιταχύνει χύνουμε τις προσπάθειες, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί κάτι τέτοιο θα χαρακτηριστεί ως κολλησιεργία. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Εμείς ε, ε, ε έχουμε εργαστεί πολύ γρήγορα, ήδη την επόμενη εβδομάδα λίγη και η προθεσμία για τις τροπολογίες. Ελπίζω να μας μιμηθεί στην ταχύτητα και το Συμβούλιο. Και συμφωνώ με τη ΣΕΡΠΑ, προσβλέπουμε σε περαιτέρω αγαστή συνεργασία με του κοιόδη ηγητέ και του λοιπού συναδέλφου και ελπίζω χάρη στη βοήθεια και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξουμε σε συμβαστικέ προτάσει. Και προσβλέπω σε ευόδοση σε των το κοινό προσπαθειών των δύο επιτροπών ΕΜΒΗ και ΕΚΟΝ. Όπω είπατε και η συζήτηση έδειξε ότι υπάρχει μεγάλο βαθμό ε, μεγάλος βαθμός σύγκλησης κοινών στοιχείων και αυτό είναι πολύ θετικό και θα συγκεντρώσουμε συγκεκριμενοποιηθεί και στην πορεία και θέλουμε συνάφεια και συνοχή μεταξύ των διαφόρων νομοθετικών προτάσεων. Πάντως μέχρι στιγμής η συνεργασία ήταν πολύ θετική και ελπίζουμε να συνεχιστεί το ίδιο επικοδομητικά. Ευχαριστώ και ο λόγος στην Πρόεδρο για να ολοκληρώσουμε. Ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την πολύ ζωηρή συζήτηση που είχαμε και για τη συμμετοχή σας που έδειξε ότι το θέμα μας ενδιαφέρει όλους και είναι και πολύ επίκαιρο. Χρονοδιάγραμμα 12 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα λίγη προθεσμία για τις ε, τροπολογίες. 22 Ιανουαρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και στην κοινή συνεδρία της Επιτροπής θα ψηφίσουμε στι 20 Φεβρουαρίου, ευελπιστώντα ότι θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου το αποτέλεσμα των εργασιών μας. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή και καλή συνέχεια.